Um, Καλησπέρα συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Να σας πω ότι τα πρακτικά τα χθεσινά είναι διαθέσιμα και εν σχολείων, τα οποία σας καλώ να κάνετε αν έχετε. Αν υπάρχουν σχόλια εγκρίνονται τα πρακτικά. Προχωράμε και πάμε σε ανακοίνωση πριν ξεκινήσουμε.